θα λάβει χώρα αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα, επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι οι παρεμβάσεις ενός λεπτού. Λαμπρινίδης πρώτα, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη είναι οι παρεμβάσει διάρκεια ενό λεπτού. Ε, έχουμε, όπω αντιλαμβάνομαι, 36 παρεμβάσει. Θα τι θα τις ε, ε, ακούσω όλε, αλλά θα με συγχωρήσετε που θα είμαι αρκετά αυστηρό με το χρόνο. Επομένω, one minute means one minute. Η πρώτη παρέμβαση είναι από τον κύριο Κουμουτσάκο για ένα λεπτό.

σε 37 διοικητικές περιφέρειες έπρεπε να απομακρυνθούν οι άνθρωποι και επίσης απομονώθηκαν πολλοί εθνικοί δρόμοι. Διαπιστώνονται ε, ζημίες κάθε μέρα. Μιλάμε για 4,5 ε, χιλιόμετρα δρόμου στο Γκαλάτσι, το οποίο επλήγει και το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πρόκειται για μια πραγματική καταστροφή. Πλήττονται 8.000 άνθρωποι και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση η κυβέρνηση. Θα πρέπει να προωθήσουμε την χρήση του Ταμείου Αλληλεγγύης μέχρι τις 15 Ιουλίου και μετά την αποτίμηση των ζημιών θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των Ρουμάνων πολιτών που επλήγησαν. Σβένσον, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτό το χρέος. Κατανοούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν από πού μπορούν να περικόψουν, δηλαδή βρίσκονται σε μία ιδιαίτερα ε, επιζήμια κατάσταση και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Το παγκόσμιο κύπελο λύγει και άρα δεν θα βλέπουμε την Αφρική κάθε μέρα. Θα ναι. πρέπει όμως να προσδώσουμε μεγάλη σημασία στην Αφρική και σε αυτούς που πεθαίνουν κάθε μέρα από πείνα και δίψα που δεν έχουν πια κανένα μέσο στη διάθεσή τους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα προβάλλουμε, στην, να την αναπτυξιακή βοήθεια. Ο κύριος Μασίπ Χιτάλγκο, για ένα λεπτό. Αυτός ο χώρος ελευθερίας μας θυμίζει τον Σαραμάγκο, ο οποίος ε, έρχεται από το Βιέδο που είναι δικιά μου η πόλη. Το Βιέδο που αν ξέραμε τι κάναμε θα το κάναμε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μην ξεχνάμε ότι αντιτάθηκε στον πόλεμο του Ιράκ, ότι ήταν υπέρ κάθε ταλαιπωρημένου, κάθε αδικημένου. Κομμουνιστής δεν σταμάτησε ποτέ να κατακρίνει τα σφάλματα του καθεστώτος της Κούβας, για παράδειγμα. Έδωσε μάχες στην Ιβηρική Χερσόνησο, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, παντού. Όλα αυτά δεν χάνονται. Ζήτω ο Χωσέ Σαραμάγκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Κοπά, για ένα λεπτό. Η Τουρκία ως υποψήφια χώρα οφείλει να συμμερίζεται τις αξίες και τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζονται στις συνθήκες. Επομένως, έχει ουσιώδη σημασία η δέσμευσή της για σχέσεις καλής γειτονίας, όπως επανειλημμένα έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αλλά μία δέσμευση που δεν σταματά στα λόγια Στι 30 Ιουνίου η Τουρκία προέβησε καινούρια προκλητική ενέργεια στη θαλάσσια περιοχή του Βορείου Αιγαίου εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδα. Το τουρκικό υδρογραφικό και ωκεανογραφικό σκάφος Τσεσμέ έπλεε 13 μίλια βόρεια τη νήσου σαμοθράκη και 10 μίλια από τι ακτέ τη θράκη, χωρί να έχει ενημερωθεί η ελληνική πλευρά για την πορεία και τι δραστηριότητε του. Η βελτίωση των διμερών σχέσεων είναι προ το συμφέρον και τη Ελλάδα και τη Τουρκία. Η ηγεσία τη Τουρκία έχει το τελευταίο διάστημα μιλήσει για νέο κλίμα στι ελληνοτουρκικέ σχέσει όμως οι συστηματικές παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου της ελλάδος από την τουρκία θέτουν αναπάντητα ερωτήματα για την ειλικρίνεια των προθέσεων. για μια ακόμα φορά από το βήμα αυτό θα ήθελα να καλέσω τα αρμόδια όργανα της ευρωπαϊκής ένωσης να στείλουν ένα σαφές και ηχηρό μήνυμα στην άγκυρα για την ανίκη αυτή συμπεριφορά. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία από τις μεγαλύτερες προόδους της ε, ε, ιατρικής είναι οι εμβολιάσεις. Χιλιάδες παιδιά έχουν καταφέρει να παραμείνουν στη ζωή και να ξεπεράσουν ασθένειες οι οποίες σε άλλες εποχές θα μπορούσε να τους κοστίσει τη ζωή. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δούμε όλες οι ασθένειες οι οποίες μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό ότι είναι απαραίτητο να δίνουμε αυτή τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αυξήσουμε το ποσοστό εμβολιασμού στον τρίτο κόσμο, ώστε ασθένειες οι οποίες έχουν εξαπλωθεί σε μεγάλο βαθμό να μπορούν να εμποδιστούν. Υπάρχει λοιπόν μια δυνατότητα με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσουμε την προσωπική ασφάλεια των παιδιών. Και αυτό βοηθάει και τις οικογένειε των παιδιών. Είναι απαραίτητο λοιπόν να καταλάβουμε ότι ο εμβολιασμό δεν ωφελεί μονάχα συγκεκριμένα παιδιά, αλλά και όλη την κοινότητα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε μια ευρύτερη διανομή των εμβολίων και των βασικών ουσιών που είναι απαραίτητε, ώστε να εξασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια και την υγιεινή του κοινού. Και αυτό πρέπει να είναι από του βασικού στόχου τη ευρωπαϊκή πολιτική υγιεινή. Ευχαριστώ. <clears throat> Ο κύριο Γκάλαχερ για ένα λεπτό. Uh, Θα ήθελα να υποστηρίξω την κυρία ε, Μαγκίνες σε σχέση με το Equitable Life και θα ήθελα να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί έτσι θα ήταν δίκαιο. Ε, έχω δεχτεί σωρία αιτημάτων από την ε, εκλογική μου περιφέρεια και θα πρέπει να δούμε και τις δημοσιονομικές προοπτικές 14 Νομίζω λοιπόν ότι με αυτή τη συνάντηση που θα γίνει την Πέμπτη θα πρέπει να προβάλλουμε και μία σωστή ΚΑΠ μετά το 2013. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι δαπάνες της ΚΑΠ αποτελούν το 0,4% του ΑΕΠ. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις, ιδιαίτερα την διατροφική ασφάλεια, το περιβάλλον, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και να, την επιβίωση των αγροτικών περιοχών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ρουμανία εδώ και μια εβδομάδα αγωνίζεται κατά των πλημμυρών που έχουν οδηγήσει σε 23 νεκρούς και πάρα πολλούς άστεγους. Μέσα στις συνθήκε αυτές ελπίζει η Ρουμανία να έχει και χρηματική υποστήριξη από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση της ε, Ρουμανίας δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ε, πλημμύρες, και να αντλήσει τα συμπεράσματα αυτέ, θέλω να κάνω μία έκκληση προ τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να υπάρξει η απαραίτητη υποστήριξη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό στην ε, Ρουμανία. Είναι απαραίτητο επίση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει και περαιτέρω το Ταμείο Αλληλεγγύη, ώστε να υπάρξει ένα σημαντικό ποσό το οποίο θα μπορεί να ανακουφίσει τι φυσικέ καταστροφέ. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη βοήθεια όλων, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Φλάσακ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα συμπεριλαμβάνουν Περιλαμβάνουν προφανώ και τους ε, καινούριου σιδηροδρόμου που έχουν προβλεφθεί, αλλά το πρόβλημα είναι ότι τελικά παραμένουν 16 χιλιόμετρα που πρέπει να περάσουν από ουδέτερη περιοχή των τσεχικών βουνών. Έχει χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα από ευρωπαϊκά ταμεία και η συγχρηματοδότηση θα χορηγηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Τσεχική Δημοκρατία Ευρωπαϊκή Δε Επιτροπή Το περασμένο Μάρτιο είχε δηλώσει στον Τσέχο Υπουργό Μεταφορών ότι η αξιολόγηση του προγράμματος έχει σταματήσει να γίνεται. Και παρακαλώ να το ξανασκεφτούν διότι το κοινό δεν είναι ικανοποιημένο με αυτή την απόφαση. Και πεθαίνει κόσμος γιατί, γιατί δεν υπάρχουν καλοί δρόμοι ούτε και ανσιδηρόδρομοι. ότι η ανεργία εκτινάσεται στα ύψη σε όλε τι χώρε τη ευρωπαϊκή ένωση όπου παίρνονται σκληρά αντιλαϊκά μέτρα. συνολικά στα κράτη μέλη τη ευρωπαϊκή ένωση έφτασε στα 23.113.000 ανέργους, ανέργου δηλαδή 1.801.000 περισσότεροι από το μάη του. 2009. στην ελλάδα εκτινάχθηκε στο 10,2% στην πραγματικότητα όμως υπερβαίνει το 15% τσακίζει το 23% των νέων και πάνω από το 27% στις νέες κοπέλες η κυβέρνηση του πασόκ κραδένει το μνημόνιο που από κοινού συνυπόγραψε με την ευρωπαϊκή ένωση το διεθνές νομισματικό ταμείο με τη στήριξη και των άλλων κομμάτων του κεφαλαίου και του ευρωμονόδρομου και προωθεί την κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αυξάνει τα όρια των ομαδικών απολύσεων περικόπτει δραματικά τις αποζημιώσεις απόλυσης και τους μισθούς των νεοεισερχόμενων νέων στην εργασία κατά 20% επεκτείνει την παιδική εργασία βαφτίζοντας την μαθητεία εντείνοντα την άγρια εκμετάλλευση των νέων. η βάρβαρη αυτή καπιταλιστική πολιτική χαρακτηρίζει την πολιτική τη ευρωπαϊκή ένωση και των αστικών κυβερνήσεων στα κράτη μέλη τη. η αντιλαϊκή πολιτική συνοδεύεται από τη συκοφάντηση και την ποινικοποίηση των αγώνων του ταξικού εργατικού κινήματο στη χώρα μα με ένα και μοναδικό στόχο να φορτώσουν τα βάρη τη καπιταλιστική κρίση στον εργαζόμενο λαό για να διασφαλίσουν τα κέρδη των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων. για τον εργαζόμενο λαό είναι επιτακτική ανάγκη η συσπήρωση και κλιμάκωση του αγώνα του για την ανατροπή τη αντιλαϊκής πολιτική για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονε ανάγκες του. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τούσα και να μου υπενθυμίσει η γραμματεία παρακαλώ να του αγοράσω ένα ρολόι. Ο κύριος Αγκουράκης για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σε μια περίοδο που όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαδίζουν στα χνάρια των πρόσφατων αντεργατικών μέτρων στην Ελλάδα, κλιμακώνονται τα αντιδημοκρατικά, αντικομουνιστικά μέτρα και προβοκάτσιες των κρατών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να καταγγείλω συγκεκριμένα την ποινικοποίηση των κομμουνιστικών συμβόλων στην Πολωνία, την ποινικοποίηση της ιστορικής αλήθειας στην Ουγγαρία που αμαυρώνει την αντιφασιστική νίκη των λαών, θα ήθελα επίση να καταγγείλω την απαγόρευση των κομμουνιστικών συμβόλων από μια κυβέρνηση προ-Ευρωπαϊκή ένωση στη μολδαβία και ανάλογα μέτρα στη ρωσία. με την ευκαιρία θα ήθελα για άλλη μια φορά να καταγγείλω την απόπειρα συκοφάντηση τη θυσία εκατομμυρίων κομμουνιστών και αντιφασιστών εξισώνοντα τον κομμουνισμό με τον φασισμό όπω πολύ καλά γνωρίζετε. οι απειλέ περί πραγματικότητα των απεργιών και των λαϊκών αγώνων δεν μπορούν να σταματήσουν την κοινωνική εξέλιξη την πάλη των εργαζομένων για την ανατροπή των βάρβαρων αντιλαϊκών μέτρων η τεράστια εκστρατεία κατά του σοσιαλισμού έχει σκοπό να πείσει τους λαούς ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. εμείς είμαστε αισιόδοξοι με σιγουριά βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη ξέρουμε ότι αυτός ο αγώνας είναι η μοναδική ε, ρεαλιστική εναλλακτική λύση στην κρίση που βιώνουν. Συνάδελφοι, σαν αντιπρόεδρος της ομάδας για τις αναπηρίες θα ήθελα να υπογραμμίσω τη μεγάλη σημασία που έχει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει στη συνειδητοποίηση από την κοινωνία των πολιτών των προβλημάτων των συνανθρώπων μας αλλά δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένες χώρες καθυστερούν γενικά τη διαδικασία. Ευχή μου είναι λοιπόν να ξεκινήσει από εδώ μια νέα όθηση έτσι ώστε να απομακρυνθούν και να ξεπεραστούν όλα αυτά τα εμπόδια, τα εμπόδια και να επικαιρώσουμε την σύμβαση αυτή των Ηνωμένων Εθνών για την Αναπηρία. αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πραγματικά να παίξει ηγετικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, δεν μπορεί να καθυστερεί και να στερεί τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν αναπηρίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυκλοφόρησε τελευταία σε ελληνική μετάφραση το βιβλίο του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Αχμέντα Βούτογλου με τίτλο «Στρατηγική Βάθος» στο βιβλίο αυτό εμφανίζεται το συνεκτικό γεωπολιτικό δόγμα της τουρκίας σαν τοπικής περιφερειακής υπερδύναμης με χώρο συμφερόντων από αδριατική μέχρι κίνα και με ιδιαίτερη έμφαση στην κύπρο βαλκάνια και αιγαίο. ιδιαίτερα για την κύπρο στη σελίδα 274 του βιβλίου αυτού αφιερώνεται ειδικό κεφάλαιο στο οποίο επισημαίνεται η γεωστρατηγική σημασία της ανεξάρτητα από το ανθρώπινο στοιχείο των κατοίκων την εθνικότητα και το θρήσκευμά τους γίνεται παράλληλα σαφής επεκτατικός πενιγμός για την ελληνική λύση ρόδου. μάλιστα επιλέξει αναφέρεται στο στρατηγικό αυτό εγχειρίδιο ότι όπως είπα, παρόλο που δεν έχουν καμία πληθυσμιακή προέκταση προς την κούβα και τα υπόλοιπα νησιά της καραϊβικής ενδιαφέρονται άμεσα για αυτά έτσι και η τουρκία είναι υποχρεωμένη από στρατηγική άποψη να ενδιαφέρεται για την κύπρο πέραν του ανθρώπινου παράγοντα. οι τάσεις να ανακτηθούν τέως ε, οθωμανικά ε, εδάφη η οποία στο βιβλίο αυτό αναφέρεται υποδηλώνει βία. βία στην ευρωπαϊκή ένωση δεν υπάρχει. πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα προς την τουρκία. Ο κύριος Ομπερμάερ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό βλέπουμε ότι η Ισπανία έχει προωθήσει το άνοιγμα νέων κεφαλαίων με την Τουρκία. Αντί να διαπραγματεύεται με την ε, Τουρκία λοιπόν για τέτοια θέματα της προσχώρησης θα πρέπει να αντιμετωπίσει ανοιχτά θέματα όπως είναι το Κυπριακό, το θέμα των Αρμενίων, τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα, η παρενόχληση και φόνη καθολικών ιερέων. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να πιεστεί η Τουρκία να προχωρήσει προς ταχύ, με ταχύτερα βήματα προς μεταρρυθμίσεις. Είναι εντυπωσιακό ότι η Άγκυρα ζητά από τη μία πλευρά να ανοίξουν νέα κεφάλαια, αλλά αρνείται να εκπληρώσει τα κριτήρια ένταξής της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνει να την πιέζει λοιπόν η Τουρκία και προωθεί μια διαδικασία ένταξης πάνω από τα κεφάλια των πολιτών και σε βάρος της θέλησής τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι συνάδελφοι. Εμφανίζομαι ενώπιόν σας σήμερα για να εκφράσω τη λύπη μου διότι βρισκόμαστε μεν στον 21ο αιώνα αλλά η ελευθεροτυπία δεν ισχύει για όλες τις χώρες μέλη. Είναι ακόμα στον καιρό της Ισπανικής Ιεράς Εξέτασης. Πώς είναι δυνατόν ένα συνταγματικό θεμελιώδες δικαίωμα όπως η ελευθερία της έκφρασης δεν γίνεται σεβαστό εκ μέρους ορισμένων κυβερνήσεων. Και μπορεί να θεωρηθεί η ελευθεροτυπία ως αδυναμία του συστήματος εθνικής λέει ασφαλείας. Τα δικαιώματα αυτά είναι αδιέρετα και αν δεν τίθεται θέμα απορρίτων πληροφοριών δεν μπορεί να υπάρξει <clears throat> ζημία της εθνικής ασφαλείας από την ελευθεροτυπία. Είναι πρόσχημα για να κλειστούν εφημερίδες ή για να επιβληθεί λογοκρισία. Μια χώρα που η κυβέρνησή της είναι η μόνη πηγή πληροφόρησης για τους πολίτες της δεν είναι πια ελεύθερη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Τσεσμέ διεξήγαγε χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς έγκριση της Ελλάδας υποθαλάσσιες έρευνες σε περιοχή που τόσο από νομικής όσο και από γεωφυσικής πλευράς ανήκει πέραν πάσης αμφιβολίας στην ελλάδα. αυτό προκάλεσε την έντονη διπλωματική αντίδραση της αθήνας. βασική αιτία αυτής της συμπεριφοράς που δημιουργεί προβλήματα στις σχέση καλής γειτονίας με κράτος μέλος είναι το γεγονός ότι η τουρκία δεν έχει υπογράψει και δεν έχει κυρώσει την σύμβαση για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. υπενθυμίζω ένα πολύ σημαντικό γεγονό η διεθνή σύμβαση για το δίκαιο τη θάλασσα είναι διεθνή συμφωνία μεικτού χαρακτήρα έχει υπογραφεί από την ευρωπαϊκή ένωση όλα τα κράτη μέλη και όλα τα υποψήφια κράτη μέλη εκτό από την τουρκία. αποτελεί λοιπόν αναπόσπαστο μέρο του κοινοτικού κεκτημένου. γι' αυτό το λόγο κάθε υποψήφια χώρα οφείλει να υιοθετήσει την unclos προκειμένου να ενταχθεί στην, ευρωπαϊκή ένωση. πρόκειται για πολύ σοβαρή προπόθεση η μη εκπλήρωσή τη από την τουρκία θα έχει αρνητικέ επιπτώσεις και στα επόμενα στάδια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και σε ειδικά κεφάλαια όπως το κεφάλαιο αλληλεία και ενέργειας. γι' αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να την ενθαρρύνει στο να την υπογράψει και να την κυρώσει τη συμφωνία αυτή. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία για ένα λεπτό. <laughs> Um, Συγγνώμη, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στη σημερινή μας συζήτηση προηγουμένως για την σημασία ας τα πω πολωνικά καλύτερα καλύτερα έλεγα λοιπόν στα αγγλικά ότι Ήθελα να μιλήσω για την πρωτοβουλία των πολιτών. Μιλήσαμε προηγουμένως γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι το θέμα δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε και αντίθετα πρέπει να το τονίσουμε. Γιατί η επικοινωνία είναι πολύ σημαντικό πράγμα και νομίζω ότι έχει αποσιωπηθεί σήμερα. Στη συνθήκη της Λισαβόνας είχαμε πει όταν τη συζητούσαμε ότι είναι πολύ σημαντικός μηχανισμός για τους πολίτες ιδιαίτερα. Αυτό που μας λείπει όμως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ακριβώς η επικοινωνία με τους πολίτες διότι δεν έχουμε αρκετή επικοινωνία μαζί τους. Τουλάχιστον όχι όσοι θα έπρεπε. Έχω ακούσει πολλούς συμπολίτε μου να παραπονούνται διότι δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία. Είναι στη διάθεσή τους. Πρέπει λοιπόν να συμπληρώσουμε τις εργασίες μας και με περισσότερη πληροφόρηση και επικοινωνία για αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών που είναι κάτι πολύ θετικό για μας και χάνουμε αυτή την ευκαιρία. Ενώ έτσι θα μπορούσαμε να πλησιάσουμε τον πολίτη περισσότερο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurostat έχει αυξηθεί η ανεργία. Έχει φτάσει το 9% στην Πορτογαλία. Υπάρχουν χώρες ακόμα με μεγαλύτερη ανεργία. Οι δραστικές περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις μαζί με την έλλειψη ρευστότητας της αγοράς μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφική κατάσταση σε ό,τι αφορά την ε, ανεργία. Χρειάζονται πραγματιστικά μέτρα. Οι χώρε συνοχή θα πρέπει να υποστηριχθούν από τα ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχο όμω θα πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε και την αναζωγόνηση μια ε, αγορά εργασία η οποία είναι αυτή τη στιγμή παγωμένη. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση σε όλα τα προγράμματα, να κατευθυνθούν οι επενδύσει προ παραγωγικού στόχου, να υπάρξει απλοποίηση των διαδικασιών χρήση των κοινοτικών ταμείων, να χρησιμοποιηθούν με ένα εύκαμπτο και ταχύ τρόπο. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει πλήρη υποστήριξη στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και να δοθούν ευκαιρίε για την πρώτη απασχόληση των νέων. Θα πρέπει να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχείρησει, γιατί αν η καθεμία από αυτέ προσλάβει ένα νέο εργαζόμενο, θα έχει σχεδόν λυθεί το πρόβλημα τη ανεργία στην Πορτογαλία. Ευχαριστώ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 οι αντιδημοκρατικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή προσπαθούν να θίξουν την ελευθερία έκφρασης και τύπου. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει ιδιαίτερα ότι υπάρχουν σημαντικές απειλές οι οποίες στρέφονται κατά των μέσων ενημέρωσης σε πολλές χώρες της Ευρώπης είτε πρόκειται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και σε επίπεδο Κομισιών υπάρχουν πραγματικά παραβιάσεις αυτής της κατεύθυνσης. Βλέπουμε να υπάρχει η περιστολή της των μέσων ενημέρωσης, υπάρχουν υποχρεώσεις οι οποίες τίθενται για να δοθούν κρατικές επιδοτήσεις και πολλές πιέσεις που ασκούνται στα μέσα ενημέρωσης. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι οι πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή είναι υπό απειλή από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε την έκθεση του κυρίου Ιβο Μπέλετ, να υπάρξει πραγματικά υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε τα κράτη-μέλη να σέβονται την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και προτείνω λοιπόν να διευρύνουμε την ε, εντολή του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή ώστε να λάβει υπόψη και την ελευθερία του τύπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κρατώντας τις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Επίτροπο. Πήρα το λόγο κύριε Επίτροπε γιατί ανησυχώ ιδιαίτερα για την αμοιβαία αναγνώριση των πανεπιστημιακών πτυχίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τις πολλαπλές συζητήσεις και την ξεκάθαρη νομοθετική ρύθμιση, ορισμένες χώρες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και αρνούνται να αναγνωρίσουν πανεπιστημιακά πτυχία. Αναφέρομαι στη Βουλγαρία. Πολλές φορές τα πτυχία από άλλες χώρες δεν γίνονται αντικείμενο αναγνώρισης αυτόματα όπως θα έπρεπε. Ζητούνται επιπλέον συμπληρωματικά έγγραφα τα οποία αξιολογούνται, εξετάζονται πέραν του πτυχίου και πέραν φυσικά του κόστους που προκαλεί σε χρόνο και σε χρήμα η διαδικασία αυτή η οποία πολλές φορές είναι αρνητική. Αυτό παραβιάζει φυσικά τα δικαιώματα και των φοιτητών αλλά και των πανεπιστημίων που έχουν εκδώσει τα διπλώματα και είναι φυσικά κατά παράβαση της οδηγίας 89 κάθετο 48. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ναι. θα ήθελα σε αυτή την παρέμβαση να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με τα θύματα των προσφάτων πληρωμών στην Ευρώπη. Θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα ποια είναι η κατάσταση στη Βόρεια Ισπανία, ιδίω στην Καταβρική, Αστούρια, Γαλλικία και χώρα των Βάσκων, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τι καταρακτόδε βροχέ που ξεπερνούν κάθε επίπεδο φυσιολογικών ε, βροχών, βροχοπτώσεων οι αρχέ πολιτική προστασία των περιοχών αυτών έχουν κάνει ό,τι μπορούν για να αντιμετωπίσουν τι ε, πλημμύρε αυτέ και να διασώσουν του πολίτε. Είναι η στιγμή να υπάρξει αξιολόγηση των ζημιών και να ζητηθούν βοήθειε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο Ταμείο Αλληλεγγύη τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι από τα καλύτερα εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τέτοιου είδου περιπτώσει. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια αποτελεσματική λοιπόν εφαρμογή τη οδηγία για τι πλημμύρε που θα μα επιτρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδου καταστάσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέμπερ είναι εδώ για ένα λεπτό. Ο κύριος Κάτσιν για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις 11 Ιουλίου θα έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που ο στρατός της Δημοκρατίας της ε, Σερβίας ε, υπό την ηγεσία του στρατηγού Μλάντιτς ε, έκανε τη μεγαλύτερη σφαγή, διέπραξε τη μεγαλύτερη σφαγή στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάνω από 8.000 άνδρες και νεότεροι έχασαν τη ζωή τους, εκτελέστηκαν ψυχρά. Μιλάμε για τα σύνορα επειδή ζούσαν ε, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Σερβία και ήταν Βόσνοι. Αυτό ήταν το μοναδικό τους έγκλημα. Πρόκειται για μια φρικτή απόπειρα εθνοτικής κάθαρσης και είναι φυσικά έγκλημα εις βάρος της ανθρωπότητας. Φυσικά και βγήκε κατά δίκη εις βάρος ε, των ενόχων και το Διεθνές Δικαστήριο το 2007 ε, ονομάτισε την πράξη αυτή σαν γενοκτονία. θα ταφούν τελικά γύρω στα 800 άτομα τα οποία ευρέθησαν τα τελευταία χρόνια να έχουν ταφεί σε ομαδικούς τάφους. Και για μια ακόμη φορά πρέπει να ζητήσουμε, τον να ζητήσουμε ο στρατηγός Μλάντιτς να συλληφθεί. Κύριε Πρόεδρε, η βελγική αστυνομία επισκέφθηκε την αρχιεπισκοπή της πόλεως Μαλίν για να κατασχέσει αρχεία. Εισέβαλε. Και η επιχείρηση κράτησε πάνω από 9 ώρες και μεταξύ των εγγράφων που κατασχέθηκαν υπήρχαν και καταθέσεις ε, πολιτών που δημοσιοποιήθηκαν. Εσυλήθησαν και δύο τάθη καρδιναλίων χωρίς κανένα λόγο παραβιάστηκαν τα θρησκευτικά δικαιώματα, οι αξίες και τα δικαιώματα του ανθρώπου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου. Όλα αυτά παραβιάστηκαν. Ζητώ λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στραφεί προς την Βαρόνη Άστον και να ζητήσει να ληφθούν μέτρα και να καταδικαστούν τα διπλωματικά επεισόδια τα οποία προκλήθηκαν από μια περίγραπτη συμπεριφορά μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος του κράτους του Βατικανού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 6 χρόνια, αυτό ήταν μια τεράστια πρόκληση τη διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ασχοληθεί πολύ με τα οικονομικά θέματα. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σα όμω σε κάτι το οποίο πολλέ φορέ λησμονούμε. Στι χώρε αυτέ έχουμε πολλέ εθνικέ μειονότητε. Δεν είναι άτομα τα οποία μετανάστευσαν σε αυτέ τι χώρε, αλλά άτομα τα οποία για ιστορικού λόγου, λόγω τη αλλαγή των συνόρων, έτυχε να βρίσκονται στις, στο έδαφο μια άλλη χώρα από τις δικιά τους. Είναι σημαντικό λοιπόν το γλωσσικό θέμα για αυτές τις μειονότητες. Οι χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλέ φορέ πιο φιλελεύθερε για του γλωσσικού του νόμου από ορισμένα δικά μα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό οι μειονότητε να μπορούν να νιώθουν άνετα στη χώρα του, όπου και να είναι αυτή η χώρα. Τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πολλά να μάθουν από υποψήφιε χώρε για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε θα πρέπει να απολαμβάνουν την ισότητα και την ίδια αξιοπρέπεια ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται και ποια είναι η εθνική του προέλευση. Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι υπήρξαν προβλήματα με υγειονομική περίθαλψη με Ευρωπαίους βουλευτές σε ξένες χώρες. Εμείς θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη μέρημνα για βουλευτές οι οποίοι έχουν ανάγκη καθημερινής φροντίδας και δεν έχουν ένα γιατρό μαζί τους ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, και κύριοι βουλευτές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι μα έχουν βοηθήσει σε επίπεδο υγείας στις δύσκολες αυτές τις στιγμές που χρειάστηκε να αντιμετωπίσω βρέθηκα σε ένα νοσοκομείο στη Σανκάη σε δύσκολε συνθήκε. Θα ευχαριστήσω λοιπόν όλου του συναδέλφους μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίω την κυρία Πλά, και σα ευχαριστώ όλου και πάλι. Ο Σικέρσκι για ένα λεπτό. Szanowni Państwo, kryzys gospodarczy dotyka wielu, wielu osób. Chcę Πρόεδρε, η κρίση έχει πλήξει πολύ κόσμο πάρα πολύ σκληρά. Σήμερα όμως θα ήθελα να περιοριστώ στις επιπτώσεις που έχει στους νέους και σε εκείνους που ζουν κάτω από το όριο της ανέχειας που, έχουν, που υπήρξαν άνεργοι για πολύ καιρό κλπ. Οι άνεργοι νέοι είναι το μεγαλύτερο τμήμα των ανέργων και μπαίνουν στην ενεργό ζωή χωρίς καμία προοπτική. Ξέρουμε ότι μια καλή μόρφωση είναι το κλειδί. Πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν στην ανάπτυξη καλύτερης παιδείας για τους νέους. Τώρα που κλείνουν εργοστάσια έχουν απολεστεί και άλλες θέσεις εργασίας. Ευτυχώς έχουμε ακόμη σχολεία και πανεπιστήμια που λειτουργούν και υπάρχουν δυνατότητες να δοθεί στους άνεργους αυτούς νέους επαγγελματική μετεκπαίδευση. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσεων και χαίρομαι ιδιαίτερα για την έκθεση της κυρίας Σιδονίας Γεντερζεύσκα που μας προετοίμασε μια έκθεση για τον προϋπολογισμό που δίνει ιδιαίτερη σημασία στους νέους. Η Ευρώπη κάποιων πολιτικών ανδρών δεν είναι η Ευρώπη των πολιτών, γιατί η Ευρώπη στην ουσία είναι εκτός παιδιάς. Δεν βοηθάμε και δεν δεχόμαστε τους εκπροσώπους των ανθρωπιστικών οργανώσεων ενώ υποδεχόμαστε ποδοσφαιριστές σαν βασιλιάδες. Υπάρχει γενικότερα ενδιαφέρον για αθλητικά γεγονότα, για μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά όχι για ε, τραγωδίες τις οποίες ε, ε, βιώνει ο κόσμος σήμερα και υπάρχουν οι προπονητές οι οποίοι δίνουν η εικόνα ανώτερου από τους ίδιους τους προέδρους του κράτους στη συγκεκριμένη περίπτωση της ε, Νοτιού Αφρικής. Υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα εργασίας, ε, προβλήματα θέρμανσης το χειμώνα και όλοι αυτοί υπάρχουν. Κύριε Σαρκοζή, εσείς δεν ασχολείστε με αυτούς και δυστυχώς για σας δεν έχουμε τις ίδιες αξίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων των πλημμυρών στη Ρουμανία. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους αυτούς οι οποίοι έχουν θυγεί από αυτά τα γεγονότα και τις φυσικές καταστροφές ότι βρισκόμαστε στο πλευρό τους. Δυστυχώς η έλλειψη προληπτικής υποδομής και η ελληματική προετοιμασία των ρουμανικών αρχών Παρά το γεγονό ότι υπήρχαν στο παρελθόν και αντίστοιχε καταστάσει, οδήγησαν σε σημαντικέ ηλικίε απώλειε και απώλεια ανθρώπινη ζωή. Όπω είπα και στην προηγούμενη Ολομέλεια, τονίζω και πάλι ότι θέλω να παροτρύνω την Κομισιόν να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα και να περιλαμβάνει προτάσεις για καλύτερη διαχείριση των ε, υδατίνων οδών και των ποταμών των κρατών μελών και επίσης να υπάρχουν και οικονομικά μέτρα για καλύτερες επενδύσεις για τη διαχείριση των ποταμών ώστε να μην επανέλθουν τέτοιες τραγικέ καταστάσεις στο μέλλον. Εξ ονόματος του Ρουμανικού λαού θέλω να ευχαριστήσω τη Γαλλία, την Εσθονία και το Βέλιο για την ταχεία του απάντηση μέσω του κοινού μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω ένα δύσκολο πρόβλημα που μας έχει συγχύσει όλους τους συναδέλφους από την περιοχή μου. Το Νοέμβριο του 2009 η Κουμβρία, που είναι τμήμα της περιοχής μου, έχει πληγεί, είχε πληγεί από πλημμύρε και χάθηκε και μία ζωή. Γι' αυτό έπρεπε να, γίνει, να ζητηθεί κάποια βοήθεια από τα διαρθρωτικά ταμεία. Δυστυχώς παρά τα 100.000 λίρες που χρειάστηκε να χορηγήσει η κυβέρνηση δεν έκανε αίτηση για αποζημίωση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Πιστεύω λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτή της περιοχής μου που χρειάστηκε να κάνουν επιδιορθώσεις πρέπει να τύχουν αποζημιώσεων και να κατηγορηθεί η κυβέρνηση για παράληψη. Οι πολύ σοβαρές πλημμύρες που έλαβαν χώρα στη Ρουμανία έχουν επηρεάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας μας, τη Ρουμανίας. Δυστυχώς 23 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ζωή τους πάνω από 18.000 άτομα εγκατέλειψαν τις αιστείε τους και πολλά σπίτια καταστράφηκαν. Ακόμα χειρότερο είναι το γεγονός ότι δεν έχει σταματήσει ακόμα η πλημμύρα. Η ρουμανική κυβέρνηση προσπαθεί να σταματήσει τα νερά, αλλά επίσης προσπαθεί να αξιολογήσει και τα, το επίπεδο των ζημιών και χρειάζεται να κάνει μια έκκληση για τη χρήση του Ταμείου Αλληλεγγύης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, οποιαδήποτε υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλύψει μόνο μέρος οικοδόμηση, αλλά θα είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα προς όλους τους πολίτες που χάσανε τα, την περιουσία τους μέσα σε λεφτά. Το να πάρουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δείξει στους Ρουμάνους ότι υπάρχει αλληλεγγύη και ενότητα στην Ευρώπη όταν υπάρχει μια κρίση. Γι' αυτό θέλω να παρακινήσω όλους τους συναδέλφους να καταδείξουν την αλληλεγγύη τους προς τη Ρουμανία και να εγκρίνουν την πρόταση οικονομικής αρρωγής μόλις ζητηθεί από τις Ρουμανικές Αρχές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Ιταλία αντιμετώπισαν δικτατορίες φασιστικού χαρακτήρα. Κυβερνήσεις οι οποίες άσκησαν μεγάλη βία και στο εσωτερικό τους και σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα η Ιταλία αντιμετωπίζει ένα μονοπόλιο στα μέσα ενημέρωσης λόγω της δράσης του Σίλβιο Μπορελουσκόνη. Στην ε, Ουγγαρία η κυβέρνηση του κυρίου Όρμπαν που υποστηρίζεται από ένα κόμμα το οποίο επίση εκπροσωπείται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσπαθεί να εξασφαλίσει και αυτό ένα μακροχρόνιο μονοπόλιο για τα μέσα ενημέρωση. Στη Ρουμανία ε, μέλη του κόμματος το οποίο ανοίξει στην ίδια οικογένεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ότι τα μαζικά μέσα ενημέρωσης είναι ευάλωτο σημείο της εθνικής ασφάλειας της Ρουμανίας. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διδαχθεί από την ιστορία της και θα πρέπει να αντιταχθεί σε αυτές τις άθλιες ενέργειες. Ευχαριστώ. E, Ευχαριστώ πολύ, κύριε έχει αναλάβει πλέον η Βελγική Προεδρία. Αντίθετα με την η Προεδρία δεν έχει παρουσιάσει τις προτεραιότητες της βασισμένες πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες απορίες. είναι σαφές ότι θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή εμφανίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι έχει πολλά προβλήματα η βελγική κυβέρνηση τα οποία θα πρέπει να λύσει αλλά υπάρχουν και στην τρέχουσα πολιτική ζωή και στην πολιτική συγκυρία και θέματα πολιτικά και θέματα φυσικών καταστροφών, σαν παράδειγμα που έφυξαν την Ανατολική Ευρώπη. Και για αυτά τα προβλήματα απαιτούνται ταχύτατες απαντήσεις και μέτρα και ελπίζω επιτέλους η Βελγική Προεδρία να είναι σε θέση να φέρει πέρα στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έσπευσαν να βοηθήσουν τις οικογένειες και τα θύματα γενικότερα αυτών που αντιμετώπισαν τις πλημμύρες. Did I, did I pronounce your name correctly, sir? Is it, is it Καλά το είπα, Grzyb. Ναι κύριε Πρόεδρε, είναι δύσκολο όνομα, το ξέρω, το ξέρω. Κύριε Πρόεδρε, στις 21 Ιουνίου της Ισημερίας η Ρωσία έκλεισε τις κάνουλες του φυσικού αερίου και μας είπε ότι μπορεί να κάνει και πρόσθετες μειώσεις των παροχών του στο φυσικό αερίο εάν οι Λευκορώσοι δεν πλήρωναν όσα χρωστούσαν. Εκείνοι όμως δήλωσαν ότι αυτό θα επηρέαζε όχι μόνο τις αγορές τους αλλά και το πέρασμα του φυσικού αερίου προς τη Δυτική Ευρώπη. Ευρώπη. Επομένως η Ρωσία προσπάθησε να ασκήσει πιέσεις για να αναγκάσει τη Λευκορωσία να σεβαστεί ορισμένες συμφωνίες και πρότυπα αυξήσεων των τιμών κτλ. ώστε να αναγκαστεί η Λευκορωσία ίσως να πουλήσει ορισμένες στρατηγικές της επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα της της Λευκορωσίας αμαυρώθηκε και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Τι θα γίνει για τον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις τι προβλέπει. Το 2009 είχε υπογραφεί ένα συμβόλαιο σχετικά με αυτό, μια συμφωνία. Επομένως, τελευταία ομιλήτρια για σήμερα, η κυρία Μαγκίνες για ένα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να χαιρετήσω τη σημερινή ανακοίνωση της Κομισιόν για την παρακολούθηση της λιανικής αγοράς. Αυτό θα οδηγήσει σε πιο δίκαιες και πιο αποτελεσματικές αγορές λιανικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το πρώτο βήμα στον δρόμο για μια πιο αποτελεσματική οικονομία, ιδίως στο λιανικό τομέα έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες να υπάρχει μια ανεξήγητη κατάσταση πολύ χαμηλών τιμών για τα αγροτικά προϊόντα σε πολλά κρατημένη, μεταξύ των οποίων και το δικό μου, ενώ συγχρόνω είναι στα ύψη οι τιμέ τροφίμων για του καταναλωτέ. Σίγουρα δεν λειτουργεί σωστά η αγορά, πολύ σωστά λέει η Κομισιόν. Είναι σημαντικό στο έγγραφο αυτό το ότι καταδεικνύεται όχι μόνο η οικονομική πτυχή της, του λιανικού εμπορίου, αλλά και ο αντίκτυπος στον καταναλωτή, στο περιβάλλον και στην κοινωνική δομή. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποβάλει τι προτάσει του μέχρι τι 10 Σεπτεμβρίου και ελπίζω δεν θα χρειαστούν 10 χρόνια για να μπορέσουμε να έχουμε δικαιοσύνη στον τομέα αλλιανικού εμπορίου. Γιατί αυτή τη στιγμή και οι παραγωγοί και οι καταναλωτέ χάνουν. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό μα φέρνει στο τέλο των παρεμβάσεων ενό λεπτού είναι η έκθεση της κυρίας ε, Τούρουνεν «Προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας». Το λόγο έχει η συγγήτρια για τέσσερα λεπτά, μετά θα έχουμε ένα catch the